Καλησπέρα σα και ε, επαναλαμβάνεται η σύνοδο. Τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση είναι στη διάθεσή σα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, αντιρρήσει. Δεν βλέπω να υπάρχουν λοιπόν ενστάσει, αντιρρήσει και εγκρίνεται λοιπόν ο